Περνάμε λοιπόν στην πρώτη ψηφοφορία. Καλωσορίζω την πρόεδρο της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Καταπολέμηση των απατών, προστασία των συμφερόντων των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη ανάγνωση, πέμπτη οδηγία, καμία ε, τροπολογία, ενιαία ψηφοφορία, ονομαστική κλήσης. Colleagues, um, on this vote, uh, there is one too many from... Η πράσινη ψήφισε ένας επιπλέον από τους πρασίνους. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Delegation. That's fine. Okay, the vote is now closed. Ωραία, πέρασε. Εγκρίνεται 56 υπέρ, 12 κατά. Μηδέν αποχές. And την κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και τώρα να ψηφίσουμε τις, τα θέματα που αφορούν τη λίμπε. Παρακαλώ τους αδέλφους ε, της άλλης επιτροπής να αποχωρήσουν ήσυχα. Ίσχα παρακαλώ οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Κόντ. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να ψηφίσουμε να ψηφίσουμε τώρα τις συνθήκες εισόδου και παραμονής ε, υπηκόων τρίτων χωρών για υψηλή ε, εξειδίκευση απασχόληση. Υπάρχουν δύο σχόλια πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Υπάρχει ένα σχόλιο για τις ε, τροπολογίες της ΕΜΠΛ με βάση το, ε, άρθρο 54 στη σελίδα 18 για τη συμβαστική 13 συγκεκριμένα. Δεν αναφέρεται ότι καλύπτεται από έναν συμβαστικό και στη σελίδα 37 μεταξύ των άλλων τροπολογιών της ΕΜΠΛ αναφέρεται ότι καταπίπτει αν εγκριθεί η συμβαστική αλλά συνδυάζεται με την ε, συμβαστική 14. Αν δεν έχετε αντίρρηση, προτείνω η έμπλε 11 να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από τη 13, τη συμβαστική και καταπίπτει εάν εγκριθεί η συμβαστική 13 ή όχι 14. Εάν το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα, καλό θα ήταν. Γιατί εντάξει είναι περίπου κατανοητό, αλλά ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία. Τροπολογία 129. Απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής. Είστε όλοι έτοιμοι. Απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής. Άρχεται. Πέρας.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 Go to Amendment 305. The vote is open. 305. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε από κοινού 3, 284 και 306. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. 307 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.36 άρχεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβαστική για το άρθρο 3. Συμβαστική 3 λοιπόν, άρχεται. Ε, ε, δική μου είναι η έκθεση. Θα πρέπει να τα ξέρω αυτά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 3.36 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 348. Άρχεται. 348. 348. Δεν έχετε ακόμη ψηφίσει όλοι. 348. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 5.2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 4-16 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 449. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 7α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστεί για το άρθρο 9. Α, συγγνώμη, όχι. Για το άρθρο 8. 8 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αλλά 10 συνάδελφοι δεν ψήφισαν. να ε, σπρώχνετε, να σπρώχνετε πιο βαθιά την ε, κάρτα σας στο μηχάνημα και να μην κοιτάτε τα τηλέφωνά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για το άρθρο 9. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι ενδιαφέρεστε, αλλά όχι τόσο πολύ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 10. Άρχεται. Άρθρο 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 13 που καλύπτει και την τροπολογία 11 της ΕΜΠΛΑ, άρχεται πέρας το EFTD έχει μια ψήφο παραπάνω. Παρακαλώ, διορθώστε το. Ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε Λοιπόν, τροπολογία 508. 508 άρχεται. 508 πέρας απορρίπτεται 509 άρχεται πέρας απορρίπτεται 507 άρχεται πέρας Απορρίπτεται. Από κοινού 5.13, 5.10 και 5.11 άρχεται. Και συμπεριλαμβάνει και την 5.14 αυτή η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτονται. Συμβαστική για το άρθρο 14 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 19 Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 569. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστή για το άρθρο 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας για το άρθρο 23 άρχεται. ΕΛΚ μία παραπάνω. Ωραία. Διορθώθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. τροπολογία 6, 25 και έμπλε 19 ταυτόσιμες άρχεται. Πέρας Εγκρίνονται. Συμβαστική για το άρθρο 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 25. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127 και 635 που είναι ταυτόσιμες άρχεται πέρας εγκρίνονται τροπολογία 636 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 128 και 637 που είναι ταυτόσιμες άρχεται Πέρας. Εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις. Αιτιολογική σκέψη 1. Συμβαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 136. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική 3α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική 3αα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της ιτολογικής 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της 4B ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, όχι, τροπολογία 139, άρχεται. 139. Άρχεται. ΕΛΚ μία παραπάνω. Παρακαλώ διορθώστε το. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της 5 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της 5 5α άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική έπιψη τιολογικής 5B. Άρχεται. Πέρας. Έλξη μία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική ε, συγγνώμη, 150. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 154. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 155. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 6α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 6b. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική της αιτιολογικής 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί αιτιολογικής 8α. Ε, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 168. Άρχεται. Πέρας. Απολύπτεται. Συμβαστική επί της 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική επί της αιτιολογικής 13. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Και παρνάμε στην αιτιολογική σκέψη 14. Δύο ψηφοφορίε 183. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 184 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για την ιδεολογική σκέψη 15. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για την ε, ιδεολογική σκέψη 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το 17 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 210 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για την σκέψη 20. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 2.14 παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 215 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για τη λογική σκέψη 21. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Για την 22, τη λογική σκέψη 22. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 223. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται σε και για τη λογική σκέψη 24. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για την ιδεολογική σκέψη 26 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για τη λογική σκέψη 27. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εντελεγική σκέψη 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Έναρξη. Πέρας. Έγκρινεται. 34α. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 35. Συμβαστική για τη λογική σκέψη 35. Ψηφίζουμε. Πέρας. Τώρα πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική για τη λογική σκέψη 36. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για 36α. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αντιλογική σκέψη 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 257 και 2... 257. Είναι ταυτόσημε οι 257 με τη 258, Τι ψηφίζουμε από κοινού λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για τη τελική σκέψη 40 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 41. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σχεδόν τελειώνουμε. 42. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 74 παρακαλώ, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 46α, συμβαστική επιτελογική σκέψη 46α. Πέρας. Εγκρίνεται. 48α. Ψηφίζουμε. Σχεδόν τελειώσαμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι δύο, συγγνώμη, η συμβαστική επί της συντελογικής σκέψης 48β, παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 279. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Επί του τροποποιημένου κειμένου ψηφίζουμε. Ονομαστική κλίση. Vote is Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 44 ψήφοι υπέρ 10 κατά 2 αποχές και να ψηφίσουμε για το επί του νομοθετικού κειμένου έναξη ψηφοφορίας για την έναξη των διαπραγματεύσεων πέρας εγκρίθηκε 44 ψήφοι υπέρ 10 κατά 3 αποχές so... Συγγνώμη που πήρε τόση ώρα η ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα να περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Φαγιών. Να ρωτήσω κατά πόσο θέλετε να πάρετε το λόγο. Τάνια, όχι, δεν επιθυμείτε το λόγο. Μπορούμε να περάσουμε παρακάτω στην ψηφοφορία. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, λίγη υπομονή παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι παίρνει πολύ ώρα αυτή η ψηφοφορία, αλλά είναι και πολύ σημαντικό το θέμα αυτό τη ψηφοφορία αυτή για τα πρόσφατα αυτά. Έχουμε την ε, τροπολογία 264 της κυρίας Πινέλη, η οποία καλύπτεται από την ε, σχετική στην ε, συμβιβασμού, αλλά η τροπολογία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ψηφοφο... της ψηφοφορίας. Αν δεν διαφωνείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Στη σελίδα 33, επίσης, η ψηφοφορία unblock για τις φυσικές, για τις καταστροφές είναι σε επιπρόσθετη με τα θέματα σοβαρών ζημιών και έχει να κάνει 33 με την 36α τη εισηγήτρια και θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στο πρώτο τμήμα τη ψηφοφορία και η 68-69 η οποία έχει να κάνει με το άρθρο που περιλαμβάνονται και θα πρέπει, δυστυχώ συνάδελφοι, να σα διαβάσω αυτά. Η 215 Καστάλντο, η οποία περιλαμβάνεται στην ψηφοφορία μπλοκ, καλύπτει τι ίδιε ιδέε αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν, θα ήθελα την 23 να τη θεωρήσουμε ότι θα ψηφιστεί στο ίδιο μπλοκ. Και τέλος, στο δεύτερο, στην δεύτερη ομάδα είναι η 2.18, η 23 είναι παρόμοια με την 2.15 και παρουσιάζεται στη δεύτερη τμήμα της, των ομάδας των, ψηφο, των τροπολογιών. Αν δεν υπάρχουν αντίρρηση, να ψηφιστεί στο πρώτο τμήμα με τον 2.15. Με τις ευκρινήσεις λοιπόν αυτές μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Uh, Και περνάμε στην 96, 97, 98, οι οποίε είναι ταυτόσιμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ε, ένας από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην συμβαστική 33. Έναρξη. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1 για το άρθρο 2, για τους ορισμούς. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 324. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η 324 από μόνη της. Πέρασα. Απορρίπτεται. Η 325 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται. Συγγνώμη, ξεχωριστή ψηφοφορία, συνάδελφοι, για το άρθρο 2.9, την εισαγωγική παράγραφος για το κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1C για την ιδεολογική σκέψη 16. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 169. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 339. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται.

Η 343 με τη 214 που είναι ταυτόσιμες, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. Συμβαστική 2 για το άρθρο 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 για το άρθρο 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 για το άρθρο 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 για το άρθρο 7. Ψηφίζουμε. Τώρα ψηφίζουμε. Πέρας. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 για το άρθρο 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 για το άρθρο 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεμιβαστική 7 για το άρθρο 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7α για την αιτιολογική σκέψη 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Σε βεβαστική 8 για το άρθρο 11 ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Συμβαστική 9 για το άρθρο 12 και λογικές σκέψεις. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 12. 7, 407-408. Ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 463 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 11 για τα άρθρα 14 και 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 για τα άρθρα 15 και 21. Ψηφίζουμε. Αν ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 για το άρθρο 16. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία μπλοκ από την 69 μέχρι και την 546 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Το ανακοίνωσε και στην αρχή της ψηφοφορίας. 69 με 546. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στη συμβιβαστική... Α, συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα της ψηφοφορίας Unblock, η 549. Παρακαλώ. Και η 218 συνάδελφοι. Δεύτερο τμήμα της ψηφοφορίας Unblock, η 549, η 218 και η 219. Το δεύτερο τμήμα της ψηφοφορίας Unblock είναι η 549 και η 219. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 13 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 573 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η ε, 575 παρακαλώ, ψηφίζουμε. Η 575. Πέρα. Πέρα στις ψηφοφορίες. 576 άρχεται η ψηφοφορία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν γίνονται καθόλου λάθη. Συμβιβαστική 16 άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, δεν έκλεισα την προηγούμενη. Δεκτή η 576. Ίσως να πηγαίνω πολύ γρήγορα. Θα επαναλάβω την τελευταία ψηφοφορία. Θέλετε να επαναλάβω την 575 και την 576. Λίγη ηρεμία παρακαλώ. Ας επαναλάβουμε λοιπόν. 575 ψηφίζεται. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίες. Απερίφθη. 576. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 16 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 17 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 18 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Μπορείτε να διορθώσετε στο τέλος την ψήφο σας. Δεκτή. Συμβιβαστική 23 άρχεται. Και 31α άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 19 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 19α άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 20 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 21 ψηφίζεται. Πέρας. Το ΕΛΚ συνένα, Πέρας. Δεκτή. 691. Ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφη. Συμβιβαστική 22 άρχεται. πέρας. Δεκτή. Συμβιβασική 24 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. δύο άρχεται. Πέρας. Sorry, that is rejected. Απερίφη. Amendment 703. The vote is open. 703. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 25. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Και χωρισμένη ψηφοφορία στο άρθρο 31.1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 26 άρχεται. Τέλος. Δεκτή. 7.33 ψηφίζεται. Πέρας. Απεριφθεί. 7.14 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 715, 716 ταυτόσημες Πέρας. Πέρας. Απερίφθη. Απερίφθησαν. 717 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 27 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 28 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 29 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 30 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 31 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 771 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 772 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 773 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 32α άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 32β άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 95 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 7.95 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 7.97 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 798 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 99 στην 4 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 100 ψηφίζεται. πέρας. Συμβιβαστική 34 στις αιτιολογικές σκέψεις πια ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 35 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 36 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 37. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 163. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 171. Άρχεται.

Τέλος. Απερίφθη. 175 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 14, 176 και 177 από κοινό ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 38. Τέλος. Δεκτή. 39. Πέρας. Δεκτή. 21 και 208 ταυτόσημες. Ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 209 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 210 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 211 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 24 και 221 ταυτόσημες. Άρχεται. Πέρας. Δεκτές. 224. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 40. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική, ή μάλλον 2.38 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 41. Άρχεται. Τέλος. Δεκτή. 2.54. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 2.56 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 42. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2.63 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 43 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2.87. Άρχεται. Πέρας. Απερίφη. 290 και 291 ταυτόσημες. Ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφη. Μετά πάμε στην τροπολογία 4. Ψηφίζεται. Αιτιολογική σκέψη 6. Τροπολογία 4. Ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 9. Ψηφίζεται την τροπολογία 9. Πέρας. Δεκτή. Πάμε στην τελική ψηφοφορία ονομαστική κλίση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. 40 υπέρ 13 κατά 4 αποχές. Τώρα απόφαση εντολής διαπραγματευτικής. Ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «37 υπέρ 14 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Φαϊόν. Τάνια θα ήθελε να μας πει κάτι, έχεις το λόγο. Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας συνεργασία, να ευχαριστήσω την Αγγέλικα, την Αλεσάνδρα, την Μπάρμπαρα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά, είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας για το άσυλο. Νομίζω είναι ένα βήμα για να γίνει το σύστημα πιο ανθρώπινο. Σας είμαι ευγνώμων. Ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολλή δουλειά κρύβεται πίσω από τις εκθέσεις αυτές. Ευχαριστούμε λοιπόν την Δάνια, ευχαριστούμε και τους Κιώδες, ευχαριστούμε και όλους τους υπαλλήλους για τη βοήθειά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, συνάδελφοι, για τις σημερινές ε, ψηφοφορίες.